Allora, buongiorno Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε. Έγκριση τη ημερήσιας διάταξη. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει, θεωρούμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Να δώσω απευθεία το λόγο στον Επίτροπο Τσιόλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα εδώ σήμερα θα μας κάνει μία ενημέρωση για την ε, κρίση σχετική με το βακτηρίδιο του Εσερίκ που όπως ε, γνωρίζουμε όλοι δυστυχώς προκάλεσε το θάνατο 38 ατόμων στην Ευρώπη και σοβαρά προβλήματα υγείας σε περίπου 3.000 άτομα. Το καλό νέο είναι ότι η πηγή της ε, μόλυνσης έχει πλέον εντοπιστεί και πλέον φαίνεται ότι έχουμε ξεπεράσει την κρίση. Όμως οι Ευρωπαίοι παραγωγοί οποροκυπευτικών πλήχθηκαν και ακόμα πλήττονται από τι συνέπειε ε, για τι υποψίε, οι οποίε αποδείχθηκαν αθασμένε, οι οποίε αποδόθηκαν σε πολλά οπορεκυθαριστικά προϊόντα. Ε, τα προϊόντα ε, ε, τα οποία δεν πουλήθηκαν ε, εκτιμώνται ότι είχαμε μια απώλεια της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ την εβδομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ισπανία και οι παραγωγοί που χτυπήθηκαν περισσότερο ήταν η Ιταλία, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Γαλλία. Ε, προβλέπονται πάνω από 210 εκατομμύρια ως ποσό για την αποζημίωση και πρέπει να θεωρηθεί αυτό το πρώτο βήμα, αλλά Φυσικά το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψουμε τις ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν. Επίσης, η κατάσταση αυτή καταδεικνύει πως η διαχείριση κρίσεων στην Ευρώπη θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω προκειμένου να ανταποκριθούμε με αποτελεσματικό και ταχύ τρόπο σε ανάλογες κρίσεις. Ε, Προσφάτω ε, μεταβήκαμε στι Ηνωμένε Πολιτείε, αγαπητοί Ντάρσιαν, και διαπιστώσαμε πόσο ένα σημαντικό τμήμα του νόμου για τη γεωργία, του Farm Bill, είναι αφαιρεωμένο ακριβώ στη διαχείριση κρίσεων. Ο Επίτροπο πρέπει να φύγει στι 10.30. Θα ήθελα να ζητήσω στου συναδέλφου να σταθούν μόνο μόνο στο θέμα των, ε, ε, του βακτηρίου Σεχίρ και τα μέτρα τα οποία λήφθησαν για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω απευθείας το λόγο στον Επίτροπο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, όπως το τονίσατε, και όπως ε, είναι πολύ γνωστό από τις 26 Μαρτίου όταν η ε, κρίση σχετικά με το βακτηρίδιο αυτό επεξετάθη στον τομέα των ε, ε, οποροκυπευτικών της Ευρώπης υπήρξε σοβαρότατη κρίση με σημαντική μείωση των πωλήσεων και των τιμών ακόμη και αν ήδη ε, πριν από μερικές εβδομάδες πριν εμφανιστεί το βακτηρίδιο του Έσεριχ υπήρχαν χαμηλότερες τιμές λόγω της συγκυρίας. Η ανάκαμψη της αγοράς θα εξαρτάται πάντοτε από την ε, εμπιστοσύνη των καταναλωτών και για να αποκατασταθεί η ε, εμπιστοσύνη έπρεπε να εξευρεθεί η πηγή της μολύνσεως. Στη Γερμανία όμως ε, μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτή την πηγή και προσπαθούμε να δούμε τα στοιχεία σχετικά με τις πωλήσει αφού ε, ενετοπίστη η αιτία της μόλυνσης για να δούμε πώς εξελίσσεται η αγορά. Από την αρχή ο στόχος μας ήταν να μπορέσουμε να επέμβουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα διότι όπως σας είπα και εγώ κάποια στιγμή ε, όχι για πολύ καιρό αλλά υπήρξα παραγωγός οπωροκυπευτικών και ξέρω τι σημαίνει ε, στην παραγωγή αυτή ένα ευρώ το οποίο ε, αποζημιώνεται εντός ε, εβδομάδων είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ένα ευρώ το οποίο αποζημιώνεται μετά από χρόνια. Γι' αυτό και το ανέφερα ή στο Συμβούλιο και καθότι η τελευταία μεταρρύθμιση της αγοράς ε, δεν έχει προχωρήσει η αγορά δεν μπορεί να αντιδράσει πάρα πολύ γρήγορα και ελπίζω ότι με την αποδοχή του νομοθετικού πακέτου που θα υποβάλουμε η Επιτροπή θα έχει τη στήριξη του Συμβουλίου και του ε, ε, ε, ε, του Κοινοβουλίου για να μπορέσει να αντιδρά γρήγορα. Με την εφαρμογή ε, αυτών των μηχανισμών της αγοράς σε τέτοιες κρίσεις δεν ε, έχουμε επαρκή μέτρα για να δράσουμε και γι' αυτό παρακολούθησα την ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για να δούμε πώς θα επηρεάσουμε και θα αναμορφώσουμε το άρθρο 190 για να μπορούμε να αντιδράσουμε και να επέμβουμε σε περιπτώσεις σαν την παρούσα. Ε, ήδη λοιπόν υπήρξε μία έκτακτη συνεδρίαση του ε, Συμβουλίου των Υπουργών επί του θέματος και ε, απεφασίστη μία αποζημίωση όλων των παραγωγών 50% για αυτούς που δεν είναι μέλη των οργανώσεων παραγωγών και φτάνοντας μέχρι 70% για τις οργανώσεις ε, των παραγωγών οι οποίες ε, ναι μεν έχουν ήδη μέσα για να προβούν σε αποζημιώσεις και ε, επιλέξαμε τα προϊόντα που είχαν επηρεαστεί περισσότερο από την κρίση λόγω της πτώσεως της εμπιστοσύνης των ε, καταναλωτών και των προϊόντων για τα οποία έχουμε ίσως ε, τεχνικά λιγότερες δυνατότητες ε, αποταμιεύσεως για ε, να ε, ε, αντιπαρέλθουμε εις την διάθεση της παραγωγής. Δηλαδή για ευαίσθητα προϊόντα όπως είναι τα αγγούρια, οι ντομάτες και τα ε, ε, ε, οι πιπεριές και τα κολοκυθάκια. Δηλαδή αυτά ήταν τα προϊόντα τα οποία είχαν πληγεί περισσότερο και γι' αυτά η δυνατότητα προσαρμογής της συγκομιδής ή τη διάθεση είχε μειωθεί σημαντικά προβλέψαμε 210 εκατομμύρια ευρώ ε, για ε, τη χρηματοδότηση αυτής της αποζημίωσης αλλά όπως είπα στην αρχή αυτή ήταν η πρώτη κινητοποίηση ε, πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο αλλά θα αναλύσουμε τις αιτήσει των μελών των παραγωγών των οργανώσεων των παραγωγών που θα υποβληθούν μέχρι τέλος Ιουνίου και θα αποσταλούν από τα κράτη-μέλη ε, αρχές ε, Ιουλίου ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναλύσουμε τα στοιχεία, να δούμε ποιες είναι οι αιτήσει, τι ποσό ζητείτε και θα μπορέσουμε έτσι να αναλύσουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε εις το φάκελο μετά από το τέλος του Ιουνίου ένα ποσό βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί. Θα αρχίσουμε να καταβάλουμε τις αποζημιώσεις τον Ιούλιο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ζήτηση και η αγορά. Έχουμε ένα πλαφόν, μία οροφή για να αποφύγουμε σε ορισμένες περιοχές υπερβολική αντιστάθμιση διότι δεν υπήρξε πάντοτε η ίδια η διακρίση σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης και υπάρχει μία περίοδος αναφοράς στην οποία έχουμε καθορίσει για τον Ιούνιο μεταξύ του 2008 έως το 2010 και θεωρείται ε, ότι ε, η βάση αυτή χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστεί η αποζημίωση και στην περίοδο αυτή αν δείτε την τιμή αναφοράς θα δείτε ότι ήταν υψηλότερη από την τιμή την οποία είχαμε εφέρει φέτος τον Ιούνιο και πριν ξεκινήσει η κρίση. Χρειάστηκε λοιπόν αυτή η περίοδος αναφοράς που έπρεπε να καθοριστεί για να έχουμε επαληθεύσιμα ε, θέματα σαν αναφορά αλλά στα περισσότερα προϊόντα θα είναι προς όφελος των παραγωγών διότι η παραγωγή ήταν ε, ήδη χαμηλότερη κατά 50% από, σε σχέση με την τωρινή ποσότητα ποσότητα και τιμή. Προ... λοιπόν ε, μία αποζημίωση και για τα μη μέλη των οργανώσεων αγοράς και επίσης ε, πήραμε μέτρα ε, για ορισμένες εξαιρέσεις, για οργανώσεις παραγωγών, για ορισμένα όρια τα οποία είχαμε προβλέψει στον κανονισμό για την απόσυρση των προϊόντων και την δυνατότητα να αποζημιώσουμε. Υπάρχει ένας περιορισμός χρηματοδότησης από το επιχειρησιακό ταμείο των οργανώσεων αυτών για τέτοιες κρίσεις που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 τρίτο του προϋπολογισμού και εξαλείψαμε όλους αυτούς τους περιορισμούς για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τις οργανώσεις των παραγωγών να μπορέσουν να ενεργήσουν χωρίς να επηρεάσουν την ε, ε, ε, συνεκτικότητα των προγραμμάτων τους μετά την κρίση. Προς το παρόν δεν έχω ακόμη τα στοιχεία για την εξέλιξη της αγοράς μετά την ανακοίνωση της κρίσεως και ε, του εντοπισμού της πηγής της μολύνσεως και ελπίζω ότι στις αρχές επομένης εβδομάδος θα έχω αυτά τα στοιχεία και θα σας τα στείλω για να μπορέσετε να παρακολουθείτε και να έχετε σημεία αναφοράς παρακολουθώντας την εξέλιξη της κρίσεως. Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητή Επίτροπε, ευχαριστώ Ντάτσιαν για αυτή την τόσο σημαντική ανακοίνωση. Να ξεκινήσουμε τώρα αμέσως τη συζήτηση. Για άλλη μια φορά θα ήθελα... Συγγνώμη. Ένα ακόμη σχόλιο διότι θα υπάρξουν ερωτήσεις πέραν αυτή της ε, αποζημιώσεως στους επόμενους μήνες θα χρειαστούν ε, ενέργειες προωθήσεως και επικοινωνίας για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην κατανάλωση των ε, οποροκυπευτικών διότι είδαμε ότι και λαχανικών ιδίω διότι δεν φταίει όλος ο τομέας ή ο συγκεκριμένος τομέας παραγωγής AUTHORWAVE και πρέπει ε, να ξεκινήσουμε μέτρα και να προσπαθήσουμε να επιταχύνει η Επιτροπή την ανάλυση για να αναλάβει μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο και ελπίζουμε ότι το φθινόπωρο θα είμαστε έτοιμοι με ορισμένα προγράμματα επικοινωνίας που θα ξεκινήσουν από το φθινόπωρο κατά τρόπον ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε τον τομέα των λαχανικών λοιπόν το δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε μέσα στη συζήτηση, να ζητήσω από τους αδέλφους να τηρήσουν τα όρια, ε, ο, ο Επίτροπος έχει μισή ώρα. Απευθείας ο Άλμπερτ Ντες. έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα εδώ και ποτού, προτού συζητήσουμε συγκεκριμένα για τα λαχανικά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πληγήκαμε από μία κρίση η οποία έχει ήδη πολύ σημαντικές επιπτώσεις και για τους ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν από αυτή ε, της, ε, ε, της μολύνσεως στη Γερμανία υπήρξαν 39 νεκροί και ένας υψηλός αριθμός ασθενών και ο Υπουργός ε, ο Ερμόδιος Υπουργός στη Γερμανία έλαβε μέτρα αλλά πάντοτε υπάρχουν επιπλήξεις και κάθε φορά που ε, ε, πεθαίνει ένας ασθενής αμέσως ο τύπος γράφει ότι είναι ανθρώπινο λάθος οπότε θέτω το ερώτημα έχουν, έχει ενημερωθεί το κοινό εγκαίρος αυτό είναι διαφοροποιημένο διότι στη Γερμανία υπάρχει ε, στο ομοσπονδιακό επίπεδο μία, ε, ε, μία διαφορετική δομή και ελέγχθη ότι οφειλόταν η μόλυνση αυτή σε ισπανικά αγγούρια. Αλλά αυτή η ενημέρωση απευθυνόταν μόνο στους Γερμανούς των βορείων κρατηδίων. Παρόλα αυτά όμως έπαυσαν όλοι να τρώνε ντομάτες και ε, δεν θέλω γι' αυτό το λόγο να ζητήσω περισσότερες αποζημιώσεις αλλά δεν επλήγησαν μόνο ορισμένα λαχανικά διότι οι καταναλωτές δεν έτρωγαν πλέον ούτε μοτσαρέλα δεν είχαν ντομάτα δεν έτρωγαν μοτσαρέλα και χρειάστηκε να περιοριστεί Στή πάρα πολύ η ε, παραγωγή της μοτσαρέλα διότι κατέρευσε το σύστημα. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για τη γρήγορη αντίδρασή σας κύριε Επίτροπε και να σας πω ότι ε, σας ευχαριστώ που το αρχικό ποσό των 150 εκατομμυρίων έφτασε στα 210 και ξέρουμε όλοι ότι δεν θα επαρκέσει για όλες τις αποζημιώσεις. Η ερώτησή μου λοιπόν κύριε Επίτροπε είναι η εξής. Μπορούμε να κάνουμε ε, προσπάθειες όλοι μαζί για να έχουμε επαρκή χρηματοδότηση να αντιμετωπίσουμε τέτοιες κρίσεις στο μέλλον και θα υπάρχουν πάντοτε κρίσεις ασχέτως της μορφής τους. Πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε, πρέπει να το συζητήσουμε με τους οικονομολόγους, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλό θα ήταν 2% των χρηματοδοτικών πόρων να μπορέσουν ετησίως να διατίθενται σε ένα ταμείο κρίσεως αφού εξασφαλιστεί ότι τα λεφτά αυτά θα παραμείνουν στο ταμείο αυτό και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους στόχους ε, για τον Γαλιλαίο ή για κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να έχουμε μία μακροπρόθεσμη προοπτική ε, συγκεντρώσεως πόρων για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις. Ευχαριστώ, Άλβερτ. Η κυρία Γκαρσία Πέρες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη σημερινή του παρουσία εδώ στην Επιτροπή προκειμένου να μας παρουσιάσει τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν για την κρίση η οποία ε, προέκυψε στον απορροκευτικό του ε, από το βακτηρίδιο ε, ΣΕΡΙΧ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι συμπάσχω με τις οικογένειες οι οποίες πλήχθησαν από το συγκεκριμένο πρόβλημα. νομίζω ότι δεν θα πρέπει να λησμονούμε και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν από το πρόβλημα και στους οποίους δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας. Θα ήθελα να δούμε και τα θέματα τα οποία πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να απαντήσουμε εμείς ε, ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τα όσα προέκυψαν από αυτή την κρίση. Στη συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, κατά την άποψή μου παρουσιάσαμε τα ζητήματα στα οποία είχαν γίνει μοιραία σφάλματα όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης. Ε, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο σε κάποιο βαθμό λειτουργήσε στην πηγή μεν, αλλά δεν αναφερθήκαμε στη διανομή και στην αντιμετώπιση και αυτό έπληξε πάρα πολύ σοβαρά όλο τον ευρωπαϊκό τομέα και ιδίως ε, τη χώρα μου την Ισπανία. Το αποτέλεσμα ήταν ε, απώλεια εσοδείας, απώλεια εισοδημάτων και δυσφήμιση για την εικόνα των γεωργών. Αυτή η απάντηση λοιπόν που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα για την επίλυση της κατάστασης μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και για τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις ακόμα και οι οποίες ε, έχουν ε, ληφθεί υπόψη από κάποια κράτη-μέλη, διότι η πρόταση κανονισμού δεν ήταν ε, ομόφωνη. Υπήρχαν τέσσερις χώρες που καταψήφισαν και κάποιες ε, χώρες οι οποίες ήταν ε, απήχαν της διαδικασίας. Ο Επίτροπος βέβαια έδειξε ότι είναι διατεθειμένος να συμπληρώσει τα πράγματα ανάλογα με το πώς ε, θα προχωρήσουν τα θέματα της κρίσης. Ε, σε αντίθεση με τα όσα συνέβησαν στο γαλακτοκομικό τομέα πριν από δύο χρόνια, δεν έγινε κατανομή των πόρων αναχώρα, το οποίο κατά την άποψή μου θα ήταν εσωτική σημασία και επιπλέον το σύστημα των αποζημιώσεων ευνοεί χώρε οι οποίε αυτή τη στιγμή ε, έχουν την ε, εσοδεία των προϊόντων τα οποία θα αποζημωθεί και δεν να λαμβάνονται υπόψη το γεγονό ότι υπήρξαν κάποιε χώρε οι οποίε επλήγησαν από την πρώτη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν κάποια συζητήματα τα οποία είναι ζωτική σημασία για να δώσουμε μια αποτελεσματική απάντηση και θα μπορούσαμε να τα λάβουμε ω συμπληρωματικά μέτρα. Οι αποζημιώσει που προβλέπονται στον κανονισμό, από ό,τι κατάλαβα, θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλα προϊόντα, να καλύψουν και άλλα φρούτα και άλλα κυπευτικά ε, εποχιακά και νομίζω ότι πέραν του κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο και να προσπαθήσει να αποφύγει οποιαδήποτε αυθαίρετη δράση των εμπορικών μας εταίρων, όπως για παράδειγμα το κλείσιμο των συνόρων χωρίς λόγο. Επιπλέον, Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια κάποια ελαστικότητα στην εφαρμογή του κανονισμού για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στις συνθήκες κάθε περιοχής. Χαίρομαι που άκουσα ε, στο τέλος της παρέμβασής σας ε, ότι υπάρχουν και κάποιες ε, εκστρατείες προώθησης. Είναι σημαντική σημασία σε αυτός, είναι σημαντικό και υπάρχει και ο κανονισμός για την προώθηση των προϊόντων μας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως μέσο για αυτό το λόγο. Είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η τιμή των ευρωπαϊκών προϊόντων και δεν νομίζω ότι, δεν θα, ότι θα πρέπει ε, να ε, παραλείψουμε να κάνουμε εκστρατείες για προώθηση των προϊόντων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα γνωστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών προϊόντων και τέλος Νομίζω ότι στη μελλοντική συζήτηση για την κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να βρούμε νέα μέσα τα οποία θα μπορέσουν να είναι πιο αποτελεσματικά για την ανταπόκριση σε κρίσεις όπως αυτή που αντιμετωπίσαμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολύ λίγα λεπτά στη διαδιάθεσή μα. Θα ζητήσω συγγνώμη στου αδέλφου. Προ το παρόν δεν έχω ε, παρέμβει στου συντονιστέ, αλλά μετά θα πρέπει να ε, περιορίσουμε το χρόνο. George Lyon. Ε, θα είμαι πολύ σύντομο. Πρώτο ερώτημα. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε τις πηγές που έχουν εντοπιστεί ή ταυτιστεί οφείλονταν το βακτηρίδιο η Οφείλω όταν το βακτηριδιο η υπαρξη του σε, σε αυτό που είπε ο τύπος ή τι δημιούργησε όλη αυτή την κρίση γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δεύτερον η αντίδραση και η δυσκολία εντοπισμού της πηγής. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι η Κομισιόν και οι άλλες αρμόδιες αρχές θα κάνουν μια διαφανή και πλήρη ανάλυση για να δούμε πού υπήρξε το λάθος, αν υπήρξε λάθος και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιωθεί στο εξή η ανταπόκριση σε τέτοιου είδους κρίσεις. Γιατί όλα αυτά έχουν τεράστιες επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και καταστράφηκαν, ζημιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό πολλοί γεωργοί και άλλοι. Και τρίτο ερώτημα. Ε, are we any closer to get... Ότι η ρωσική αγορά θέλουμε να ανοίξει και να λειτουργεί με τις μεθόδους του ελευθέρου εμπορίου, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο και να ανοίξει και η ρωσική αγορά στην Ευρώπη πρέπει να υπάρχουν τέτοιες διαφανείς διαδικασίες. Τέλος, μήπως στον προϋπολογισμό μπορεί να γίνει κάτι για να αντιμετωπίζονται τέτοιες κρίσεις. Μάρτιν Όσλιν. Ναι κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Η κρίση ακόμη δεν έχει περάσει. Έχουμε και νέους ασθενείς ή στην ε, ε, Γερμανία. Δεν αναφέρομαι εδώ στις επικεφαλίδες των νέων, αλλά απλούστατα πρέπει να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε από πού προέρχεται αυτή η μόλυνση που δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής. Ε, ε, τίθεται λοιπόν ερώτημα στη Γερμανία τουλάχιστον για το τι πρόκειται να συμβεί ακόμη με την κρίση αυτή και τι μας περιμένει. Δεν πρέπει λοιπόν να μιλάμε μόνο για αποζημίωσεις και να θεωρήσουμε ότι τα άλλα θέματα είναι λελιμένα. Πρέπει να σκεφτούμε και τις αιτίες αυτής της κρίσεως, δηλαδή από πού προέρχεται και σας υπενθυμίζω ότι έγινε μία μεγάλη συζήτηση για τη χρήση των αντιβιωτικών ή στην ε, κτηνοτροφία και ε, είδαμε ότι οι επιπτώσεις ε, της ασθενείας με τα δυσκολία αντιμετωπίζονται, οι επιπλοκές της ασθενείας, οπότε ε, πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε γιατί άργησε να εφαρμοστεί ο μηχανισμός κρίσεως, διότι η Ευρώπη και πάλι χρειάζεται ένα καλύτερο τρόπο διαχειρίσεως των κρίσεων. Λέγεται ότι δεν τα έβγαλε πέρα καλά και όσον αφορά την, ε, τις αρμοδιότητες των υγειονομικών αρχών και των ε, αρχών ελέγχου η αντίδραση άργησε και δεν ήταν κατάλληλη και σωστή. Χρειάζεται λοιπόν ευρωπαϊκό συντονισμό σε τέτοιες κρίσεις κατά τρόπον ώστε να λέμε ότι υπάρχει μία αποτελεσματική και αξιόπιστη αντίδραση και μπορούμε να γνωρίζουμε ε, πώς και αν χρειάζεται να αλλάξουμε τις διατροφικές μας ε, συνήθειες, τις καταναλωτικές μας συνήθειες ε, και πώς αυτό επηρεάζει τις δομές. Πρέπει τελικά να θέσουμε το θέμα ενός ταμείου κρίσεως, διότι από πού προέρχονται τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται, αυτό είναι ένα ερώτημα και επιπλέον πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν ε, κάθε φορά να θεωρούμε ότι μπορούμε να ε, ε, να ικανοποιήσουμε και να αποζημιώσουμε όλες τις ζημίες διότι αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες δηλαδή η μη κατανάλωση ενός ε, υλικού ε, ε, ενός τροφίμου σημαίνει ότι καταναλώθηκε κάτι άλλο επίσης πρέπει να δούμε πόσο θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί λαχανικών και τέλος, ε, ολοκληρώνω ρωτώντας πώς θα φροντίσετε στο μέλλον εφόσον αυτή δεν είναι η τελευταία κρίση θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ε, έναν ε, μηχανισμό και προειδοποίησεως και αποζημιώσεως στην Ευρώπη για να μην υπάρχει το χάος το οποίο διαπιστώσαμε τις τελευταίες εβδομάδες στην Ευρώπη. James Nicholson. Και εγώ θα είμαι συντομότατος. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς όσους υπέφεραν ή πέθαναν, ή τις οικογένειες αυτών που πέθαναν από αυτή την κρίση, καθώς και των παραγωγών που υπέστησαν ζημίες. Είναι προφανές ότι άμεσες αντιδράσεις και δηλώσεις μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλο κακό. Πρέπει να βασιζόμαστε πρώτα στα γεγονότα. Πράγμα που δεν συνέβη κατά την πρώτη φάση της αντίδρασης. Τα σημαντικότερα έχουν τεθεί βέβαια ήδη όπως είπαν και προηγούμενοι ομιλητές. Η ανάλυση που πρέπει να κάνετε πρέπει να καταλήξει σε μαθήματα σε διδάγματα. Γιατί συνήθως ξεχνάμε τα προηγούμενα. Υπήρξαν και άλλες κρίσεις που επηρέασαν ολόκληρη την Ευρώπη. Και ορισμένες από αυτές δεν περιορίζονται στα σύνορα μίας χώρας. Είστε ικανοποιημένος, θεωρείτε ότι η Ένωση έχει τον τρόπο να ανταποκριθεί σε τέτοια και ανάλογα προβλήματα ή κρίσεις. Ότι δηλαδή υπάρχει ο μηχανισμός που απαιτείται. Ωραία, ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε με τους συντονιστές. Ε, τώρα αγαπητοί συναδέλφοι σας παρακαλώ να... Λορέντσο, θέλεις το λόγο, συγγνώμη δεν σε είχα δει. Και κατόπιν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα κι εγώ. Ένα σημαντικό ζήτημα κύριε Επίτροπε είναι το εξή. Νομίζω ότι πριν από κάποιου μήνε ε, διαπιστώνουμε ότι για του γεωργού υπάρχουν πάντα κρίσει. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή μέθοδο για να παράγουμε και από πλευρά μέσων ενημέρωση, ε, που όπω είπατε και εσεί είναι σημαντικό, διότι διαπιστώνουμε ότι τελικώ αυτοί που ε, πλήττονται είναι παραγωγή. Δεύτερο σημαντικό θέμα είναι τα κονδύλια τα οποία δίνονται τώρα, όπως είπε ο Πρόεδρος προηγουμένως, πρέπει να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα μόνο, γιατί η κατάσταση είναι πολύ σοβαρό και πρώτοι θα να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσουν στους παραγωγούς και ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα από τη διάθεση των κονδυλίων μέχρι την άφηξή τους στους παραγωγούς που είναι αυτοί οι οποίοι πάσχουν από αυτή την κατάσταση. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά την άποψή μου σε αυτές τις δύο πτυχές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Εγώ σε ευχαριστώ Λορέντσο. Η κυρία Ραντς Καρσία για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μπω κατευθείαν στην ουσία. 39 νεκλούς και όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έχασαν τις ε, ε, θέσεις εργασία τους ε, για αυτή την κρίση από το αγκουράκι και νομίζω ότι ε, η κατάσταση είναι πολύ σημαντική. Μπορεί να δημιουργηθούν ε, πολλά προβλήματα από οποιοδήποτε Ευρωπαίο πολίτη και θα πρέπει να δοθεί ιδέουσα πωλήση. 250 εκατομμύρια ευρώ είναι ψυχία σε σχέση με αυτό το οποίο προκλήθηκε. Δεν υπήρχε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης κινητοποίησης τις κρίση ε, σε διατροφικά θέματα. Ε, υπάρχουν ένα δις ευρώ το 2011 τα οποία δεν διατίθεκαν και εσείς δίνετε μόνο 250 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την κρίση η οποία προέκυψε και από κακό χειρισμό της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπή. Δεν καλύπτονται τα προϊόντα και η παραγωγή με ισότιμο τρόπο και δεν καλύπτονται όλοι οι παραγωγοί σε μεγάλες ζημίες πρέπει να δίνονται μεγάλες βοήθειες και δεν συνέβη αυτό αυτή τη στιγμή. Είχαμε μεγάλες ζημίες και τους δίνουμε ψίχουλα για να αποκαταστήσουμε την εικόνα των ε, ισπανικών προϊόντων τα οποία ε, χάθηκαν πρέπει να εργαστούμε το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Γιατί πρέπει να περάσει το καλοκαίρι και να δράσουμε τον Οκτώβριο, γιατί πρέπει να περάσουν αυτοί οι μήνες, πρέπει να αποκαταστήσουμε το συντομότερο δυνατόν την ε, εικόνα η οποία πλήχθηκε που δεν έχει σχέση μόνο με τους Ισπανούς, Πορτογάλους, Γάλλους, Ιταλούς παραγωγούς, με όλους τους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος να σας πω ότι ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να παρουσιάζονται βιολογικά γκουράκια στην ε, κατάλογο ε, και θεωρείται ε, προϊόν το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο. Φαίνεται ότι δεν έχει αφαιρεθεί από τη λύση και η απάντηση είναι ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Σας παρακαλώ βάλτε τους υπαλλήλους σας να εργαστούν και θα πρέπει να εξαφανιστούν όλες οι αναφορές και να μην υπάρχει το προϊόν στον κατάλογο αυτό. Ζητώ συγγνώμη συναδελφοί, αλλά είναι μετρημένα τα λεφτά που έχουμε στη διάθεσή μας και πρέπει να απαντήσει ο Επίτροπος, ο Ζωζέ Μποβέ. très vite. Γρήγορα, σύντομα και εγώ. Τρία ερωτήματα. Πρώτον, για τον προϋπολογισμό και το Ταμείο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Πώς γίνεται να μην βρίσκουμε χρήματα ενώ στον προϋπολογισμό του 10 450 εκατομμύρια που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τη Γεωργία πρέπει να επαναδιατεθούν για το σχέδιο ΙΤΕΡ. Αυτό το βρίσκω απαράδεκτο και νομίζω ότι πρέπει να, να θεωρήσουμε αυτή την απόφαση γιατί σημαίνει ότι όταν παρατηρείται ένα πρόβλημα έλλειψη ισορροπίας δεν βρίσκεται λύση. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να πάνε σε ένα απόθεμα για τη διαχείριση των κρίσεων. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεύτερον, ο προϋπολογισμός. Φαίνεται ότι χρειάζεται καθαρά χωριστός προϋπολογισμός για την ΚΑΠ. Αληθινός προϋπολογισμός για την ΚΑΠ και να γίνουν προσπάθειες βέβαια και σε άλλους τομείς. Εγώ είμαι υπέρ της αύξησης του προπολογισμού για την ΕΦΣΑ και όλους τους οργανισμούς αξιολόγησης και ανάλυσης γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά αν δούμε τι συμβαίνει στις Ηνωμένε Πολιτείε ως προς τη διαχείριση κρίσεων σε σύγκριση με την Ευρώπη. Εμείς είμαστε σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Τρίτον και τελευταίον υπάρχει και νέο κρούσμα στη Γαλλία με τον Κιμά που επολύθη από τα καταστήματα Λίντολ στο βορρά της Γαλλίας. Πάλι με το ίδιο βακτηρίδιο. Και φαίνεται από όλα αυτά τα προβλήματα ότι δεν υπάρχει χνηλασιμότητα. Κρέατα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και που μεταφέρονται σε άλλη χώρα από τη χώρα σφαγής για την μεταποίηση τελικά δεν έχουν να αφήνουν κανένα ίχνος. Πώς μπορούμε να ταυτίσουμε την πηγή. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε το κοιμά για να δούμε από πού ακριβώς προήλθε. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχει κανένα δυνατότητα ειχνηλασιμότητας. Ατράω νεβέσου. Κύριε Πρόεδρε, Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για τα νέα τα οποία μας παρουσιάσατε και τα οποία ε, καλύπτουν τις τρεις ανησυχίες που θα ήθελα να αναφέρω και εγώ. Καταρχάς, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα οπορεκυπευτικά προϊόντα, ιδίω τα προϊόντα της Νότιας Ευρώπης. Για το συγκεκριμένο θέμα, με ικανοποιούν όλα όσα άκουσα από τον Επίτροπο και όσα, όπως και η κυρία Ερεάνς, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα, διότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στα προϊόντα αυτά. Ιδάλλως, ε, ε, λησμονούμε το γεγονός ότι η κρίση αυτή ε, είναι κρίση δημόσιας υγείας και επειδή έγινε κακοδιαχείριση της κρίσης μετατράπηκε σε πρόβλημα προκυπευτικών. Δεύτερον, οι αποζημιώσεις. Χαίρομαι που προβλέπονται περαιτέρω αποζημιώσεις, παρά το γεγονός ότι φοβάμαι ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των ζημιών που προκλήθηκαν. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα με το συγκεκριμένο θέμα της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τρίτον να αναφέρω και το ε, πρόβλημα με τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Ε, το είπε και ο Επίτροπος, θα ήθελα να μας πει κάποια επιπλέον πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει για την ε, επανεξέταση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για θέματα διαχείρισης κρίσης στο παρόν πλαίσιο της κοινή αγροτικής πολιτικής για το 2020. Ε, Κύριε Ρώτης. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι οι ενέργειες που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν επαρκούν διότι ο τομέας των λαχανικών είναι πολύ περίπλοκος και η παραγωγή είναι σε πολύ δυσχερή θέση. Επιπλέον οι ε, κινήσεις οι οποίες ανελεύθησαν είναι, ε, περιλαμβάνουν πολύ γραφειοκρατία και προσπαθούν τελικά να ικανοποιήσουν τις ε, οργανώσεις παραγωγών που δεν είναι πολύ ανεπτυγμένες ιδίως στα νέα κράτη-μέλη και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αποσμιωθούν περισσότερο η μεμονωμένη παραγωγή χρησιμοποιώντας βεβαίως τη σωστή διαδικασία θα πρέπει να υπάρξουν εθνικοί φάκελοι και να δοθούν περισσότερες δυνατότητες να υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις για συγκεκριμένες χώρες. Τα, δεν καλύπτονται όλες οι χώρες από αυτά τα μέτρα. Παραδείγματος χάρη είναι τα μανιτάρια. Είναι ένας ε, τομέας ο οποίος επηρεάζει ιδιαίτερα την Πολωνία. Όσον αφορά τη Ρωσία θα πρέπει ε, να συμπεράνουμε από αυτό το πρόβλημα ότι ε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα πρέπει δηλαδή να συζητήσουμε ε, τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ρωσίας και να εξετάσουμε και τα συστήματα ελέγχου των εισαγωγών. Η κυρία Ρόντους, ευχαριστώ για την παρουσία σας κύριε Επίτροπε, είμαστε σε μια πολύ δυσχερή κατάσταση με πολλούς θανάτους και θα υπάρξουν και άλλοι ε, εκατοντάδες ε, ασθενείς οι οποίοι είναι στην εντατική παρακολούθηση και ε, επιπλέον κάθε μέρα υπάρχουν περισσότερα κρούσματα. Φαίνεται ότι τώρα το βακτηρίδιο πέραν των φύτρων εμφανίστηκε και στο οικολογικό σύστημα, στο νερό ποταμών και έχουμε πληγή. Πρέπει να συζητήσουμε για τους γεωργούς οι οποίοι καλλιεργούν λαχανικά και οι οποίοι υπέστησαν μεγάλη οικονομική ζημία διότι ε, στη Γερμανία αυτή τη στιγμή αποφεύγουν την κατανάλωση νοπών λαχανικών. Δεν ε, πρέπει να αποζημιωθούν όσοι αποδεδειγμένα έχουν ζημιωθεί ασχέτως του είδους της παραγωγής, παραδείγματος χάρη ε, οι φράουλες ή η ρόκα η οποία δεν ε, είναι εξορισμού λαχανικό στην Ευρώπη δεν θα αποζημιωθεί ε, και λέγεται επίσης ότι θα αποζημιωθούν μόνο οι συνεταιρισμοί. Τι θα γίνει με τους παραγωγούς που δεν συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς. Μη σκεφτόμαστε ε, μόνο εθνικά, νομίζω πρέπει να σκεφτούμε ευρωπαϊκά, διότι δηλαδή θα πρέπει ε, όλοι να επέμβουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Ντές που πρότεινε ε, το ταμείο. Το είχαμε ζητήσει αυτό ήδη στην κρίση της διοξίνης και σίγουρα πρέπει να επιταχυνθεί η κατάρτισή του διότι θα υπάρξουν και επόμενες κρίσεις στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ την Κομισιόν καταρχήν για την ε, ταχεία της ανταπόκριση και χρησιμοποίηση του Ειδικού Ταμείου. Θα έπρεπε βέβαια μέσα σε δύο μέρες να πάτε και στη Ρωσία για να δείτε τι φρονούν και εκείνοι, ο συνάδελφός σας Ντάλι ιδίω. Εσείς βέβαια είστε με τη γεωργία και η δική σας ανταπόκριση ήταν άμεση. Σας ευχαριστώ λοιπόν Νομίζω ότι δεν δαπανάτε το ποσό που θα έπρεπε για τέτοια αντιμετώπιση. Αν και έχουμε 800 εκατομμύρια περίπου στο περιθώριο, ενώ χρησιμοποιούμε μόνο 210 περίπου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που ρώτησαν και προηγούμενοι, τι περιθώριο υπάρχει για καλύτερη χρησιμοποίηση του ειδικού αυτού ταμείου. Παραδείγματος χάρη οι ντομάτες και τα αγκουράκια που αποδείχτηκε ότι δεν έφταιγαν αλλά πουλήθηκαν με πολύ χαμηλή τιμή ένα-δύο λεπτά το κιλό. Οι παραγωγοί τους δεν πήραν καμία αποζημίωση. Δεν θα έπρεπε μέσω ενός συμπληρωματικού σχεδίου και αυτοί να αποζημιωθούν. Θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση παρακαλώ. Μάτω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι εκφράζω τον ελεγγύο με στα θύματα και να πω ότι υπήρξαν προβλήματα για τους ε, παραγωγούς ε, της Ευρώπης εν γέννη και για τους Ισπανούς πιο συγκεκριμένα. Και όλα αυτά χωρίς αποδείξεις, ε, χωρίς να ληφθεί ιδέουσα προσοχή. Υπάρχουν σημαντικές απώλειες, έκλεισαν αγορές και φυσικά είναι και θέμα κύρους. Παρόλο που εμείς στην Ισπανία παράγουμε με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και εγώ θεωρώ ότι στην Ισπανία παράγουμε με περισσότερα μάτρα ασφαλή δυσκολίε παγκοσμίω. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια απάντηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε αντίστοιχα θέματα να μην επαναληφθούν και να υπάρχουν και κυρώσει αν κρυθεί απαραίτητο. Χαίρομαι για τα όσα είπε ο επίτροπο, αλλά τα 210 εκατομμύρια ευρώ δεν επαρκούν. Είναι περιορισμένη η ποσότητα και είναι περιορισμένα και τα προϊόντα στα οποία απευθύνονται. Θεωρώ ότι ε, δεν θα πρέπει να έρθετε μετά να μας πείτε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα τα κονδύλια, διότι πραγματικά θα υπήρχε μικρή ε, χρήση, όχι γιατί δεν υπήρχε ζήτηση, αλλά γιατί περιορίστηκε η ζήτηση σε πολύ προϊόντα. Ο κύριος Ολενίτσκα και μετά ο κύριος Ανιό. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι σήμερα τα θέματα επιθεώρησης ε, ασφάλειας των προϊόντων ε, για τα κρέατα και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες λειτουργούν αποτελεσματικά. Υπάρχουν όμως άλλες επιθεωρήσεις που δεν λειτουργούν αποτελεσματικά. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στις διάφορες χώρες και η παραγωγή έχει ανέβει σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως στο μέλλον θα πρέπει να αναλύσουμε το σύστημα και να εξεύρουμε σύγχρονες λύσεις που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Όχι μόνο όσον αφορά την παραγωγή κρέατος ή γαλακτοκομικών, αλλά σήμερα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και το γεγονός ότι υπάρχουν απειλέ ε, και από άλλου τομεί όπως η παραγωγή απορροκυπευτικών. Αυτό ήταν το πρώτο ζήτημα. Δεύτερον, το εμπάργκο της Ρωσίας ε, δεν έχει αρθεί ακόμα και δεν υπάρχει ακόμα δυνατότητα να πολιθούν απορρεκυπευτικά και φρούτα από την Πολωνία στη Ρωσία. Οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές και αυτό είναι αποτέλεσμα συστημάτων που δεν λειτουργήσαν αποτελεσματικά. Οι έλεγχοι δεν έγιναν όπως έπρεπε και τις συνέπειες ε, τις βιώνουν οι παραγωγοί μανιτεριών όπως ανέφερε και, σήμερα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, γι' αυτό λοιπόν και κάνω έκκληση στον Επίτροπο να συμπεριλάβει και τα μανιτάρια στον κατάλογο ε, των αποζημιώσεων. Πρόκειται για άμεση συνέπεια της κρίσης και αν δεν υπήρχε η κρίση και την ε, κακή, ε, τον κακό χειρισμό της κατάστασης από τις γερμανικές αρχές, οι ε, πολωνοί παραγωγοί δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα. Ένα τελευταίο ζήτημα είναι το θέμα του εμπορίου με τη Ρωσία. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στους Γερμανούς πολίτες οι οποίοι επλήχθησαν. Κάποιοι ε, θα κάνουν και ε, Ταμείο τεχνητό νεφρό μέχρι το τέλος της ζωής τους ε, ως συνέπεια της κρίσης και θεωρώ ότι είναι πολύ δυσανάλογες οι αποζημιώσεις που ε, δόθηκαν. Θα ήθελα ο Επίτροπος να με διαβεβαιώσει ότι ε, θα πρέπει να ληφθούν, δοθούν αποζημιώσει. αποζημιώσεις. ε, θα υπάρχουν απώλειες για τη Βρετανική Γεωργία ο Τζοβάνι Λαβία και μετά ο Σέρβιο Σιλβέστρη. Ευχαριστώ τον Επίτροπο γιατί έλαβε πολύ έγκαιρα δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να το θέσω κάποιες ερωτήσεις. Γνωρίζετε ότι οι ερωτήσεις για τις ε, δράσεις ε, προώθησης ε, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά θα μπορούν να παρουσιαστούν από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Όσον αφορά την ε, τριτογενή αγορά, η προθεσμία είναι 30 Μαΐου του 2012. Επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτές οι προθεσμίες, μήπως τα προγράμματα θα πρέπει να εγκριθούν έγκαιρα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ αργά για να ανταποκριθούν στα προβλήματα της αγοράς. Δεύτερη πτυχή. Κατά πάσα πιθανότητα, σε αυτόν τον κανονισμό που έχουμε, για τη διανομή των προϊόντων θα έπρεπε να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ του προϊόντος που είναι ε, στην Ήπεθρο και των προϊόντων θερμοκηπίου. Διότι ε, για τα προϊόντα θερμοκηπίου ε, η μέγιστη ποσότητα των 300 τόνων είναι ανεπαρκής για τα προϊόντα θερμοκηπίου. Επίσης αναφέρουμε ε, σήμερα πολύ κακή χρήση για τα προγράμματα για τους ε, πιο ευάλωτες ομάδες και ε, τους δίνονται με απόφαση δικαστηρίου 113 εκατομμύρια ευρώ. Κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούσαμε να βρούμε λοιπόν και κάποιους επιπλέους πόρους και σε άλλες γραμμές προϋπολογισμού. Ο Σέργιο Σιλβέρτης, ε, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την έγκαιρη και αποτελεσματική δράση σας. Τρεις πολύ γρήγορες ερωτήσεις για τις αποζημιώσεις μας είπατε ότι έχουμε φτάσει σε ένα μέγιστο 50% σε σχέση με τις απώλειες τις οποίες διαπιστώνεται ότι έγιναν. Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι παρά το γεγονός ότι κάνει μια μεγάλη προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονίζει εργασίες για πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αυτή η κρίση αγοράς σημαίνει κίνδυνος πτώχευσης και να αποζημιώσουμε μόνο κατά 50% τις ζημίες μπορεί να μην επαρκεί για να βοηθήσουμε τους παραγωγούς και να βοηθήσουμε στην επιβίωσή τους, ιδίως τους όπου οι γεωργικέ εκμεταλλεύσεις είναι μικρές και κατακαιρματισμένε. Όσον αφορά τα εμπορικά μέτρα, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα πιστοποίησης για τις αποστολές προ τη Ρωσία που θα είναι απλό και δεν θα είναι δαπανηρό και θα μπορέσουμε να νομιμοποιήσουμε όλες τις εξαγωγέ τη Ευρωπαϊκής Ένωση προ τη Ρωσία ενώ ε, στην πράξη ήταν πολύ τοπική η αιστεία της μόλυνσης, ε, επλήχθησαν όλα τα προϊόντα. Επίσης, το γεγονός ότι έχουμε εποχιακά προϊόντα και είναι αδιανόητο να σκεφτούμε ότι θα προγραμματίσουμε σήμερα μία εκστρατεία ενημέρωση για υλοποίηση σε κάποιου μήνες. Θα πρέπει ήδη από το καλοκαίρι οι καταναλωτές να μπορούν να καθησυχαστούν και να είναι βέβαιοι ότι μπορούν να καταναλώσουν απορροκυπευτικά και φρούτα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Γκουτιέρεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις πολύ σύντομες παρατηρήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η αντίδραση ενώπιον της κρίσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διαχείριση της κρίσης και τα ότι μέλη γενέστε. Καταρχάς, πραγματικά θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έλαβε πολιτικές πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο. Δεν υπήρχε και θεσμικό συντονισμός για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Ε, υπήρχε έλλειψη συντονισμού μεταξύ των γερμανικών αρχών, των ευρωπαϊκών αρχών και άλλων των χωρών και όλα αυτά προκάλεσαν μεγάλη ανασφάλεια στους πολίτες και μεγάλη ανασφάλεια και μεγάλες απώλειες για τους παραγωγούς. Η διαχείριση της κρίσης ήταν κακή, χείριστη θα μπορούσα να πω. Ε, στα θέματα διαχείριση της κρίσης παρουσιάζονται ε, ένας κανονισμός ο οποίος δεν ήταν ομόφωνος ε, στα μέλη του Συμβουλίου ο οποίος δίνει ανεπαρκείς ποσότητες, δεν αποζημιώνει τους ε, παραγωγούς, ιδίως τους Ισπανούς παραγωγούς ε, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, δεν περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα, ε, είναι ανεπαρκή τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται, λείπουν ε, οπορεκυπευτικά, λείπουν εποχιακά προϊόντα και Επίση, κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι ο κανονισμό είναι πάρα πολύ αυστηρό. Υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και φαίνεται ότι η γραφειοκρατία δίνει την αίσθηση ότι η γραφειοκρατία θέλει να στερήσει δικαιώματα ε, αποζημίωση στου παραγωγού και τους γεωργούς μας. Σας ζητώ λοιπόν και νομίζω ότι είναι και το λογικό την ίδια ταχύτητα που δράσατε για να εγκρίνετε τον κανονισμό αυτή την εβδομάδα, θα πρέπει να κάνετε και με την ίδια ταχύτητα μια εκστρατεία προώθηση των ευρωπαϊκών προϊόντων για την ποιότητά του, ε, γιατί ε, ακόμα προλαβαίνουμε να ρυθμίσουμε ε, τα θέματα για τα οποροκυπευτικά και τα φρούτα του καλοκαιριού η μεγαλύτερη ευθύνη μας είναι να διορθώσουμε και να ε, τροποποιήσουμε όσα πρέπει να τροποποιήσουμε για τη διαχείριση αυτή της κρίσης και όλα όσα προέκυψαν από αυτή την κρίση να μην επαναληφθούν. Ευχαριστώ τον Σέρζιο, ευχαριστώ όλους εσάς, αγαπητέ Επίτροπε. Κάναμε μια απόπειρα να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι, αλλά προφανώς το ζήτημα ε, απαιτεί και την παρέμβαση όλων των συναδέλφους. Ε, έχει το λόγο, Ντάτσιαν. Είναι προφανές ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα ευρωπαϊκά οπορεκυπευτικά και φρούτα και νομίζω ότι αυτή θα είναι και η πιο άμεση δράση που μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αγαπητέ Ντάτσιαν, έχει το λόγο. Ε, ε, ότι έγινε, στην τελευταία παρέμβαση λέτε, ότι έγινε πολύ κακή διαχείριση από την Κομισιόν με μεγάλη καθυστέρηση και πολύ γραφειοκρατία. Ε, πέστε μου τότε, σε ποια πρόσφατη κρίση η Κομισιόν παρενέβη τόσο γρήγορα. Ή ανομάστε μου έναν τομέα όπου η Κομισιόν να μην έχει περιμείνει καν το τέλος της κρίσης για να παρέμβει. Δέχομαι μεν τις επικρίσεις, ιδίως όταν είναι επικοδομητικές, αλλά να λέτε ότι η Κομισιόν δεν αντέδρασε ταχαίως ή εγκαίρως, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να το λέτε σωστό. Θέλω να διαχωρίσω την αντίδραση της Κομισιόν και το τι μπορεί να κάνει για υγειονομικά θέματα και προστασία των καταναλωτών από τη μία και το θέμα της προστασίας των παραγωγών από το άλλο. Για το δικό μου θέμα μπορώ να σας απαντήσω και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το θέμα του ελέγχου της συνέχειας που θα δοθεί για το υγειονομικό πρόβλημα για αυτό το θέμα είμαι σε επαφή όπως πάντοτε με τον Επίτροπο Νταλή και παρακολουθούμε, παρακολουθήσαμε την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών ζητήσαμε ανάλυση όλων των δυνατοτήτων που υπάρχουν για αντίδραση και παρέμβαση της Κομισιόν σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά γνωρίζετε κι εσείς ότι δεν διαθέτει η Κομισιόν ε, επιθεωρητές, αλλά τα κράτη-μέλη. Εμείς έχουμε κανονισμούς και λέτε ότι είναι και υπερβολικά πολύ, Αλλά εδώ το πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός των κανονισμών, αλλά ο συντονισμός από τα κράτη-μέλη μεταξύ των δικών τους υπηρεσιών. Ξέρω ότι η Κομισιόν πρέπει να ακολουθεί, να παρακολουθεί ίσως λίγο πιο προσεκτικά και σαφέστερα πού υπάρχουν τα προβλήματα για να ξέρουμε ότι υπάρχει πλήρης διαφάνεια στο συντονισμό. Αλλά δεν κάνουμε εμείς το συντονισμό στη θέση των χωρών μελών. Αλλιώς θα χρειαζόταν να δημιουργήσουμε παράλληλες δομές με τα κράτη-μέλη. Λέτε δεν αντέδρασε η Κομισιόν εγκαίρως αρκετά γρήγορα. Εγώ δεν ξέρω αν μπορούσαμε να είχαμε αντιδράσει γρηγορότερα. Λέτε ότι δεν συντονιστήκαμε με το Συμβούλιο. Εγώ πήγα στο Συμβούλιο, στο έκτακτο Συμβούλιο με πρόταση. Αρχές Ιουνίου. Δεν περίμενα να μου πούν οι Υπουργοί ή οποιοδήποτε άλλος πρέπει να κάνετε κάτι κύριε Επίτροπε. Δεν περίμενα εβδομάδες και μέρες. Ίσως στο παρελθόν γίνονταν τέτοια πράγματα σε άλλες κρίσεις. Εγώ πήγα στους Υπουργούς με πρόταση. Η πρόταση αυτή ήταν κανονισμού της Κομισιόν και όχι του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο διαβουλεύτηκε με τα κράτη-μέλη και δεν χρειάστηκε εκεί ψηφοφορία. Ήταν κανονισμός της Επιτροπής. Γιατί αν δείτε τι κανονισμούς, τι αποφάσισε το Συμβούλιο δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε περισσότερα εργαλεία για να μπορεί το Συμβούλιο να δημιουργήσει το νομικό υπόβαθρο που να επιτρέπει στην Κομισιόν να δράσει. Εδώ όμως επρόκειτο για κανονισμό της Επιτροπής και η οποία αντέδρασε όπως έπρεπε. Για να δω τώρα ότι είναι πιο μεγάλη γραφειοκρατία. Σε μερικούς μήνες θα πάω πάλι στην Κοκομπού για να δικαιολογήσω πώς θα πανώνται τα χρήματα. Και νομίζω ότι συμφέρον όλων είναι να φανεί ότι γίνεται καλή διαχείριση. Αλλά μπορώ να σας πω ήδη ότι εμεί ζητήσαμε το ελάχιστο να περάσει από τις οργανώσεις των παραγωγών το θέμα των μέτρων που θα περνούν από δωρεάν παροχές. Αυτό για να είναι πιο ελαστική η οργάνωση της λειτουργίας των οργανώσεων των παραγωγών, αλλά δεν μπορούμε να πληρώνουμε και για προϊόντα που δεν ξέρουμε αν έχουν αποσυρθεί ή όχι ή καταστραφεί, γιατί μετά θα τεθεί πρόβλημα αξιοπιστίας του συστήματός μας. Η Κομισιόν λοιπόν πρέπει να εξισορροπήσει από τη μία την ταχύτητα αντίδρασης και από την άλλη τις αποδείξεις για τη δράση της. Έχω τους κανονισμούς εδώ και να μου πείτε ποιο είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό στοιχείο. Εμείς το ελάχιστο ζητήσαμε. Μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα εγκρίθηκε ο κανονισμός μετά την υποβολή της πρότασης. Από τη στιγμή που εγκρίθηκε λοιπόν, από τις 18 Ιουνίου, τα κράτη-μέλη μπορούν να υποβάλουν αιτήματα, να δεχτούν αιτήματα των παραγωγών και με βάση τα αιτήματα αυτά, εφόσον αποδείξει ο παραγωγός ότι καταστράφηκε η παραγωγή του ή αποσύρθηκε, Τότε τα κράτη-μέλη υποβάλλουν στην Κομισιόν τα στοιχεία και η Κομισιόν κάνει τους υπολογισμούς και αποζημιώνει. Δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω. Για τον προϋπολογισμό. Έχω ήδη πει ότι βάσει των στοιχείων μας, αν και περιμένω ακόμη να δω τα αιτήματα των χωρών μελών, βάσει των στοιχείων της υπηρεσίας μου, για τα προϊόντα που στοχεύσαμε. Σας εξηγώ ποια ήταν αυτά που είχαν επηρεαστεί περισσότερο και που ήταν τα δυσκολότερα για συντήρηση, για αργότερη πώληση. Βασιστήκαμε στις ποσότητες που είχαν παραχθεί και που δεν είχαν ακόμη πωληθεί. ...200 περίπου εκατομμύρια καλύπτουν αυτά τα προϊόντα. Σύμφωνα επαναλαμβάνω με τους υπολογισμούς που κάναμε αρχές Ιουνίου όταν δεν είχε ακόμη τελειώσει η κρίση αυτή. Γι' αυτό λέω ότι ρεαλιστικό, τους ρεαλιστικότερους υπολογισμούς θα έχουμε τέλη Ιουνίου μετά από τα αιτήματα των χωρών μελών οπότε θα ξανασυζητηθεί στη Διαχειριστική Επιτροπή το θέμα. Παρόλα αυτά προτίμησα να δράσουμε αμέσως όπως είπε και ο κύριος Νίκολσον όχι βιαστικά αλλά ταχαίως. Βασιστήκαμε στα στοιχεία που είχαμε για να έχουμε κάποια αντίδραση. Και αυτό θα χτενιστεί στο μέλλον και θα διορθωθεί με βάση τα όρια που έχουμε τον προϋπολογισμό. Δεν είπα ότι τα 200 εκατομμύρια είναι απόλυτο όριο και δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Νομίζω ότι μπορούν να ξεπεραστούν, αν χρειαστεί. Αυτό όμως θα φανεί τέλη Ιουνίου. Μην ξεχνάτε όμως, το υπενθυμίζω και πάλι, οι οργανώσεις των παραγωγών έχουν ήδη διαθέτουν ορισμένα μέσα, όχι απεριόριστα βέβαια, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από αυτές, αλλά διαθέτουν ορισμένα μέσα και δυνατότητες αντίδρασης. Ο κύριος Σεκριάτσι νομίζω είχε πει, δεν ξέρω αν έχει φύγει τώρα, είχε πει, είχε ρωτήσει γιατί οι οργανώσει των παραγωγών να ανακατεύονται εδώ και όχι με μονομένη παραγωγή. Ασχοληθήκαμε και με μεμονωμένους παραγωγούς, αλλά τα οποροκυπευτικά είναι θέμα στο οποίο η κοινή οργάνωση της αγοράς βασίζεται στις οργανώσεις των παραγωγών, γιατί θεωρήσαμε, μαζί με τους συνομοθέτες, εσάς, ότι ο καλύτερος τρόπος αντίδρασης είναι η οργάνωση των παραγωγών. Δεν ξέρω αν τώρα θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να αποθαρρυνθούν οι οργανώσεις των παραγωγών. Γιατί αυτές είναι οι ικανότερες να αντιδράσουν, οι οργανωμένοι παραγωγοί. Πρέπει να τηρήσουμε την έννοια των αναλογιών, να ενθαρρύνουμε τους παραγωγούς να οργανώνονται. Στις οργανώσεις παραγωγών λοιπόν θελήσαμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την περίοδο υποβολής των προσφορών. Τώρα, τα σχέδια, προγράμματα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τέλη Οκτωβρίου αρχικά προβλεπόταν και είπαμε ότι τα σχέδια των χωρών μελών μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 15 Αυγούστου από οργανώσεις παραγωγών κτλ. Τα κράτη-μέλη μετά θα τα υποβάλουν στην Κομισιόν για επιλογή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα μπορέσουμε να υπογράψουμε τις πρώτες αποζημιώσεις. Νομίζω ότι τα μειώσαμε σε έξι μήνες είναι το ελάχιστο δυνατόν. Δεν μπορούμε να πάμε πολύ γρηγορότερα ενώ παράλληλα να σεβόμαστε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Για την Ρωσία και τις εξαγωγές. Λίγες μέρες μετά το ξέσπασμα της κρίσης ή μάλλον μετά την ταύτιση της πηγής της μόλυνσης υπήρχε διάσκεψη Ένωσης Ρωσίας στη Ρωσία και το πρώτο θέμα που έθεσε ο πρόεδρος Μπαρόσο με τον πρόεδρο Μετβέντεφ ήταν ακριβώς το θέμα της απαγόρευσης εισαγωγών λαχανικών από την ε, προέλευση Ένωσης από τη Ρωσία, εκ μέρους της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρόεδρος της Ρωσίας το συζήτησαν. Δυστυχώς για μας σε τεχνικό επίπεδο η Ρωσία δεν αντέδρασε τόσο γρήγορα. Δηλαδή αυτά που είχαν συμφωνήσει οι δύο πρόεδροι δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί. Επανήλθε η Κομισιόν μετά στο αίτημά της και αυτή τη στιγμή σήμερα ο Επίτροπος Ντάλι με εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Εμπορίου και ΣΑΝΚΟ ακόμη ασχολείται με το θέμα πέρα από τις άδειε και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται, η Κομισιόν θεωρεί ότι η Ρωσία αντέδρασε δυσανάλογα. Γιατί είχε ήδη ταυτιστεί και ήταν περιορισμένη η πηγή της μόλυνσης σε μία περιοχή της Γερμανίας, ενώ η Ρωσία απαγόρευσε τις εισαγωγές από ολόκληρη την Ένωση. Πολύ σύντομα όμως νομίζω θα λυθεί και αυτό. Τώρα, γιατί δεν υπήρξαν ταμεία αναχώρα. Ομόφωνα οι χώρες μέλη δέχτηκαν την πρόταση της Επιτροπής, επαναλαμβάνω, δεν ήταν του Συμβουλίου. Γιατί δεν έγινε κατανομή αναχώρα, γιατί, γιατί θελήσαμε να αντιδράσουμε γρήγορα. Οποιοδήποτε πρόσθετο κριτήριο θα πρόσθεται καθυστέρηση και γραφειοκρατία. Και θελήσαμε να μειώσουμε στο ελάχιστο τα απαραίτητα στοιχεία που έπρεπε να ληφθούν υπόψη για την αποζημίωση. Η κατανομή αναχώρα, εξάλλου, δεν ξέρω αν θα ήταν και πολύ αποτελεσματική. Σα είπα ότι στα τέλη Ιουνίου, ανάλογα με τα αιτήματα που θα έχουν υποβληθεί, θα προσπαθήσω να ξαναδώ πόσα χρήματα θα χρειαστούν για τις αποζημιώσεις. Ούτως ή άλλως οι αποζημιώσεις θα είναι αναλογικές. Δεν θελήσαμε να εφαρμόσουμε το σύστημα του όποιος έρθει πρώτος για να είναι πιο δίκαια τα πράγματα και γι' αυτό περιμένουμε τα τέλη Ιουνίου να έχουν κατατεθεί όλα τα αιτήματα και μετά να αναλύσουμε πόσα χρήματα θα χρειαστούν για τις αποζημιώσεις ανάλογα με ε, τις ανάγκες των χωρών μελών. ερωτήματα για την σαφή ταύτιση της πηγής, διαφάνεια. Όπως σας είπα, υπάρχει μόνιμη συνεννόηση με τον Επίτροπο Ντάλι, ώστε ο καθένας από τους δυο μας να κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του μέσα στην Κομισιόν. Από τις πληροφορίες που έχω, η πηγή της μόλυνσης στη Γερμανία ταυτίστηκε και ο αριθμός των κρουσμάτων μειώνεται συνέχεια. Χρειάζεται κάποια βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης. Ο Επίτροπος Ντάλι ξέρω ότι στο τελευταίο έκτακτο συμβούλιο ανέλαβε τη δέσμευση να επανέλθει με περισσότερα στοιχεία και προτάσεις για να γίνονται τέτοιου είδους ταυτίσεις γρηγορότερα και γρηγορότερο συντονισμός επίσης. Πέρα από το υγειονομικό θέμα όμως που θα το αναφέρει ο Επίτροπος Ντάλι σε μερικές εβδομάδες με προτάσεις όπως είπα, το θέμα της διαχείρισης των αγορών και της διαχείρισης κρίσεων που έχουν επιπτώσει στις αγορές νομίζω ότι είναι θέμα που στο μέλλον πρέπει να διαθέτει περισσότερα κονδύλια για άμεση αντιμετώπιση και για τις οργανώσεις των παραγωγών γιατί νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να τονίζουμε τη σημασία τους. Όσο πιο οργανωμένη είναι η παραγωγή, τόσο ευκολότερα μπορούμε και εμείς να τους βοηθήσουμε και με μικρότερο κόστος. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι οργανώσεις των παραγωγών θα παίρνουν υπόψη τους και αυτοί περισσότερο στον προϋπολογισμό τους τη διαχείριση τέτοιων κρίσεων, την πιθανότητα διαχείριση τέτοιων κρίσεων, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν προβλέψει και αυτοί καμία τέτοια κρίση και γι' αυτό στα κράτη-μέλη άργησε η αντιμετώπιση γιατί χρειάστηκε στο πόδι να τα προβλέψουν όλα ξαφνικά την αντιμετώπιση δηλαδή τέτοιων κρίσεων. Δεν είχαν σχετική νομοθεσία και χρειάστηκε να την δημιουργήσουν εκ του μηδενός. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε τα εργαλεία που διαθέτουμε και από τις οργανώσεις των παραγωγών για να αντιμετωπίζουν τις κρίσεις και να, να αποφεύγεται η μείωση των εισοδημάτων. Αλλά και σφαιρικά, ενωσιακά, δηλαδή στον προσεχή κανονισμό πρέπει να υπάρχουν σαφέστερα μέτρα για να ταυτίζεται πιο σαφώς και στον προϋπολογισμό τι χρησιμοποιείται γιατί. Αν δεν έχουμε καμία τέτοια βάση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα χρειάστηκε να παίξουμε με τη, τα νομικά υπόβαθρα που είχαμε διαθέσιμα. Εδώ μπορεί να υπάρξει λοιπόν κάποια βελτίωση στο μέλλον. Για τα μανιτάρια και άλλα προϊόντα σας είπα ότι αντιδράσαμε ως προς τα προϊόντα που είχαν τη μεγαλύτερη επίπτωση. Στην αρχή προτείναμε τρία, μετά με τα στοιχεία που είχαμε είδαμε ότι υπήρχαν και τα κολοκυθάκια και οι πιπεριές που κινδύνευαν να καταστραφούν και χρειάστηκε να αντιδράσουμε και για αυτά. Για άλλα προϊόντα δεν ξέρω μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά λόγω της υπάρχουσας νομικής βάσης δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Με τον προϋπολογισμό που έχουμε. Για τη ρόκα και άλλες σαλάτες δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες τώρα για τη γλιστρίδα. Θα ταυτίσουμε όλα τα προϊόντα όπου χρειάζεται κάποια αντίδραση. Κύριε Νίκολσον, τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε. Για μένα υπάρχουν μαθήματα, ιδιαίτερα ως προς τα εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων και σφαιρικά για όλους τους τομείς και ειδικότερα για τα οποκροκυπεφουτικά μέσω των οργανώσεων παραγωγών. Για την προώθηση σας είπα, δεν περιμένουμε, μειώσαμε όσο δυνατόν περισσότερο την περίοδο υπάρχει βάση, υπάρχουν κανόνες, οι οργανώσεις των παραγωγών έχουν τη δυνατότητα με τα λειτουργικά τους προγράμματα να κάνουν και αυτές ορισμένα πράγματα. Αν το έχουν προβλέψει βέβαια. Αλλά ξέρω ότι δεν αρκεί δεν μια συγκεκριμένη επίγουσα δράση αλλά κάτι πιο σταθερό στα λειτουργικά προγράμματα των οργανώσεων των παραγωγών πιο ευρείες καμπάνιες χρηματοδότησης και για τις προωθήσεις και γι' αυτό μειώσαμε την περίοδο επιλογής των προγραμμάτων ή σχεδίων όσο το δυνατόν περισσότερο. Για τις επιθεωρήσεις ότι δεν λειτουργούν λέει επαρκώς έχω απαντήσει. Ο Επίτροπος Ντάλι θα έρθει να υποβάλει προτάσεις για να διασφαλιστεί καλύτερο συντονισμός μεταξύ χωρών μελών και σε κάθε κράτος μέλος, αλλά οι επιθεωρήσεις δεν είναι ενωσιακές, είναι εθνικές, με βάση ενωσιακούς κανονισμούς βέβαια. Για τη Ρωσία τα είπα. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα τα ερωτήματα ή τουλάχιστον στα περισσότερα. Αν έχω ξεχάσει τίποτε, να μου το πείτε. Χρειάστηκα όλο αυτό το χρόνο, νόμιζα ότι, θεώρησα ότι ήταν απαραίτητο. Πώς? Για το κρέας, δεν έχω για το κρέας κανένα στοιχείο από τον Επίτροπο Ντάλι για να μπορώ να κρίνω αν αν και πώς υπήρξε επίπτωση. Δεν έχουμε στοιχεία που να δείχνουν ότι υπήρξε επίπτωση στην αγορά, στις πωλήσει κρεάτων δηλαδή. Ίσως ακουστεί κάτι μετά, αργότερα. Α, το παρακολουθούμε και αυτό. Όσον αφορά όμως την ΕΦΣΑ ή την, τον υγειονομικό έλεγχο νομίζω ότι σε μερικές εβδομάδες ο Επίτροπος Ντάλι το επαναλαμβάνω θα έρθει με προτάσεις γιατί ανέλαβε αυτή τη δέσμευση ενώπιον του Συμβουλίου και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου λίγο πριν το έκτακτο Συμβούλιο είχε αναλάβει τέτοια δέσμευση και εκείνος θα έχει περισσότερα στοιχεία ελπίζω. Για μένα για τη λειτουργία των αγορών δηλαδή υπάρχουν ακόμη λήψεις και βελτιώσεις δυνατές. Ευχαριστώ Ντάτσιν για τις παρατηρήσεις και τις απαντήσεις σου. Νομίζω ότι σήμερα είναι πλέον σαφέστερη κατάσταση. Βεβαίως ανησυχούμε όλοι και θέλουμε να παρακολουθήσουμε τα ζητήματα αυτά και ελπίζουμε να μπορέσει να δώσει τις πλέον κατάλληλες απαντήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαίρως. Και πάλι σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Δυστυχώς υπερβήκαμε τις προβλέψεις. Ένα λεπτό διακοπή και κατόπιν θα συνεχίσουμε αμέσως. Riprendiamo i lavori. Riprendiamo il trabaco. Συνεχίζουμε τις εργασίες παρακαλώ. Passiamo al punto 4. Να περάσουμε στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης. Σημείο 4. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης ε, της Δευτέρας Μαΐου και της 11 και 12ης Απριλίου. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εκκρίνονται ε, μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Ένα λεπτό την προσοχή σας. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου στην αμοιβαία απολευθέρωση των γεωργικών προϊόντων και των αλλιευτικών προϊόντων είναι η 24η Ιουνίου 12 το μεσημέρι. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου για την απελευθέρωση των αλλιευτικών και γεωργικών προϊόντων, ξαναλέω, 24 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Ο εισηγητής ε, καλεί την Επιτροπή Ίντα να προτείνει το Κοινοβούλιο να αρνηθεί την έγκρισή του για την ε, σύναψη της συμφωνίας. Όσοι διαφωνούν με τη θέση του εισηγητή, επομένως είναι υπέρ της συμφωνίας με το Μαρόκο, θα πρέπει να καταθέσουν τροπολογία η οποία θα πρέπει να ψηφιστεί πρώτη. Εάν απορριφθεί ε, η τροπολογία θα ψηφίσουμε την πρόταση του εισηγητή. Αν απορριφθεί και αυτή δεν θα υπάρξει γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας ε, προς την Επιτροπή Ίντα. Ο πρόεδρο τη Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, ο Βιτάλ Μορέιρα, με ενημέρωσε επίση ότι η Επιτροπή θα κάνει σήμερα μια συνοδρία συγκεκρισμένων των θυρών, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει δύο πρόσφατες ε, ε, μελέτες αντικτύπτου που θα αφορούν τις συμφωνίες του Μερκοσούρ. Η συνεδρίαση προβλέπεται ως σημείο 30 της ημερήσιας διάταξης ε, της Επιτροπής ΕΝΤΕ και θα συζητηθεί το ζήτημα στις 5.30 περίπου. Όσοι ενδιαφέρονται από την Επιτροπή Γεωργίας ε, μπορούν να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Επαναλαμβάνω λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει την παρουσίαση των μελετών αντικτύπου που θα γίνει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επιτροπή ΙΝΤΑ, ε, μπορεί να πάει στις 5.30 περίπου στην ε, παρουσίαση. Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής ε, Βιτάλ Μορέιρα, πολύ ευγενικό εκ μέρους του, μπορούμε λοιπόν να συμμετέχουμε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Τώρα, ε, δεν ξέρω αν έχετε όλοι τις κάρτες σας, θα ψηφίσουμε και ο υποφαινόμενος φυσικά που δεν έχει την κάρτα του. Η δικιά μου που είναι, δεν έχω κάρτα. Δεν έχω κάρτα. Ο πρόεδρος ήρθε χωρίς κάρτα ψήφου, βοήθεια. Όχι, όχι, δεν την έχω ξετάσει στη Νέα Υόρκη, δεν την έφερα. Τέλος πάντων, θα στείλω να τη φέρουνε, στο μεταξύ μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ξεκινάμε λοιπόν συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα. Ε, η Ράτσε Γκαρσία Πέρες είναι η συγγήτρια. Θα ψηφίσουμε σήμερα λοιπόν την έκθεση της κυρίας Γκαρσία Πέρες ε, για τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα. Πρόκειται για μία από τις δύο εκθέσεις ε, για τη δέσμη ποιότητας και να σας υπενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε τους κανόνες εμπορία στην έκτακτη συνεδρίαση του Στρασβούργου στις 4 Ιουλίου. Σήμερα λοιπόν ψηφίζουμε μόνο το πρώτο τμήμα του πακέτου για τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται και για τους κανόνες εμπορία θα ψηφίσουμε ε, στο Στρασβούργο. Παρουσιάστηκαν ε, πάνω από 200 τροπολογίες στη σχετική έκθεση, αλλά χάρη στην εξαιρετική δουλειά της εισηγήτριας και των σχεδόν εισηγητών καταφέραμε να τι περιορίσουμε σε 19 συμβιβαστικές τροπολογίες. Επομένως ευχαριστώ και την εισηγήτρια και όλους τους κοιόδης εισηγητές. Σα υπενθυμίζω ότι πρόκειται για το πρώτο σημαντικό νομοθετικό κείμενο που πρέπει να εγκρίνει η Επιτροπή μα ε, μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα και γι' αυτό θα δώσουμε και εντολή στην εισηγήτρια να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο εν ώψη μιας πιθανής συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν από τη σημερινή ψηφοφορία να προκύψει σαφώ η βούληση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για τα θέματα ε, πολιτικής ποιότητας. Δεν ξέρω αν θέλετε να λάβετε το λόγο κυρία Γκαρθία Πέρε, πριν από την ψηφοφορία ψηφοφορία. Όχι, θα λάβει το λόγο μετά. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. E- Ξεκινάμε λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρθρο 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 67. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 68. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Sì, approvato. Dichiaro aperta la votazione. Εγκρίνεται λοιπόν η 68. Άρχεται η ψηφοφορία για την 69. 69. Ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορία, εγκρίνεται η 69. Και τώρα ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβασική τροπολογία 1. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Άρθρο 14. Συγγνώμη, τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία για τη 14. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 15. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Άρχεται η ψηφοφορία για την ε, υπαριθμών 2. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβιβαστική τροπολογία 3. Πέραση ψηφοφορίας για τη συμβαστική τροπολογία 3. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 82. 82 πέρασε ψηφοφορίες για την 82 εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. βασική τροπολογία υπαριθμών 4, πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 18. Πέραση της ψηφοφορίας, εγκρίνεται νομίζω. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 5. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 94. Άρχεται η ψηφοφορία για την 94. 94, πέραση της ψηφοφορίας, απορρίπτεται νομίζω, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 97. Άρχεται η ψηφοφορία για την 97. Πέρασε ψηφοφορία ψηφοφορίας για την 97 απορρίπτεται. «96. Άρχεται η ψηφοφορία. 96. αρχεται η ψηφοφορια 96 Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Άρχεται η ψηφοφορία για την 100. Πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται νομίζω. Τροπολογία 99. Άρχεται η ψηφοφορία για την 99. Πέρασε η ψηφοφορία για την 99. Απορρίπτεται. 101. Άρχεται η ψηφοφορία για την 101. Πέρας της ψηφοφορίας για την 101 εγκρίνεται. Εκατόν δύο. Άρχεται η ψηφοφορία για την 102. Πέρασε ψηφοφορία ψηφοφορίας για την 102 εγκρίνεται. 103. Άρχεται η ψηφοφορία για την 103. Πέρασε η ψηφοφορία για την 103. Υπήρξε ένα πρόβλημα από πλευρά τη εισηγήτρια εδώ, λέει ο πρόεδρο. 105. Ψηφίζουμε την 105. Άρχεται η ψηφοφορία για την 105. Πέραση ψηφοφορία ψηφοφορίας για την 105 εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τις ψηφοφορίας εγκρίνεται. 107. Άρχεται η ψηφορία για την 107. Πέραση της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 21. Άρχεται η ψηφοφορία για την 21. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 108. Άρχεται η ψηφοφορία για την 108. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα η τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 109. Άρχεται η ψηφοφορία για την 109. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 110. Άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι, πέρασε της ψηφοφορία για την 110, εγκρίνεται. 113. Άρχεται την ψηφοφορία για την 113. Πέρασε της ψηφοφορία για την 113. 114. Εγκρίθηκε η 113. Άρχεται η ψηφοφορία για την 114. Πέρασε η ψηφοφορία για την 114. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 115. 115. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία για την 115. Εγκρίνεται. 116. Άρχεται η ψηφοφορία για την 116. Πέρας τη ψηφοφορίας εγκρίνεται. 118. Άρχεται η ψηφοφορία για την 118. Πέραση τη ψηφοφορίας για την 118. Εγκρίνεται. 119. Άρχεται η ψηφοφορία για την 119. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 120. Άρχεται η ψηφοφορία για την 120. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 121. Άρχεται η ψηφοφορία για την 121. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 122. Άρχεται η ψηφοφορία για την 122. Πέρασε της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την 123. Ψήφισαν όλοι για την 123. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 6. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 6. Ψήφισαν όλοι. Πέραση τη ψηφοφορίας εγκρίνεται. 129. Ψηφίζουμε την 129. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 24. Άρχεται η ψηφοφορία για την 24. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 7. Πέρασε τις ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβιβαστική τροπολογία 8. Πέραση ψηφοφορία Εγκρίνεται. 138. Άρχεται η ψηφοφορία. Καλώς, εγκρίνεται η 138. 140. Άρχεται η ψηφοφορία για την 140. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 140. 141. Άρχεται η ψηφοφορία για την 141. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 143 είναι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της 143. Πέρας της ψηφοφορίας. Πρώτο τμήμα της 143 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το δεύτερο τμήμα της 143. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. 144. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 145 τώρα. Πέραση ψηφοφορίας για την 145. Εγκρίνεται. 148. Άρχεται η ψηφοφορία για την 148. Πέραση τη ψηφοφορίας για την 148 εγκρίνεται. Και τέλος, 149. Άρχεται η ψηφοφορία για την 149. Πέρασε η ψηφοφορία για την 149. Εγκρίνεται 149. Πάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 9. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία τη εισηγήτρια υπαριθμών 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. εγκρίνεται. Εκατόν Άρχεται η ψηφοφορία για την 158. Πέρασε η ψηφοφορία για την 158. Απορρίπτεται. 160. Άρχεται η ψηφοφορία για την 160. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 29 της εισηγήτριας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 161. Άρχεται η ψηφοφορία για την 161. Πέρας τη ψηφοφορία Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 12. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 166. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία για την 166. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13. 13. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 13. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 της εισηγήτριας. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της Εγκρίνεται. 178. Άρχεται η ψηφοφορία για την 178. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 179 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το δεύτερο τμήμα. Ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε για το δεύτερο τμήμα καταπίπτη. 32. Κλείνει η ψηφοφορία, ενεκρίθη. Τώρα έχουμε τη συμβιβαστική 14 προς ψήφιση, ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία, εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 15, ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ενεκρίθη. Η ε, τροπολογία 186 ξεκινά η ψηφοφορία σχετικά με την 186. Ψηφίσατε όλοι, λίγοι, απερίφθη. 34 του εισηγητή για την 34 ε, του εισηγητή, λίγη ψηφοφορία, ενεκρίθη. Συμβιβαστική 16. Ψηφίσατε όλοι, λίγη. Η συμβιβαστική 6, 16 ε, ενεκρίθη. Τώρα ψηφίζουμε την 197. Παρακαλώ να συγκεντρωθείτε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ο Μάρκ Ταραμπέλα έχει ψηφίσει. Εντάξει. Λίγη ψηφοφορία ενεκρίθη. Και τώρα πάμε, πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. 198. Λίγη ψηφοφορία στην 198. Ενεκρίθη. 199 ξεκινάει η ψηφοφορία για την 199. Λίγη. Ενεκρίθη νομίζω. 201. 201 ε, ξεκινάει η ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία, Απερίφθη. 202. Ψηφίζουμε τη 202. Ξεκινά. Λίγη. Ενεκρίθη. Τροπολογία 203. Ξεκινάει ψηφορία για τη 203. Λίγη. Ενεκρίθη. 204 Παπαστάμκος. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι για τη 204, ενεκρίθη. 205, ξεκινά η ψηφοφορία για τη 205, λίγη η ψηφοφορία, ενεκρίθη. 206. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τη 206. Λίγη. Ενεκρίθη. 207. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τη 207. Λίγη. Ενεκρίθη. 208. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τη 208. Λίγη ενεκρίθη. Συμβιβαστική 17. Η συμβιβαστική 17 ξεκινάει ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία, ενεκρίθη. Τώρα ψηφίζουμε την 228 στην επόμενη σελίδα. Λίγη ψηφοφορία, ενεκρίθη. 230. Ξεκινάει η ψηφοφορία για 230, Ντόρφμαν και η λοιπή. Λίγη. Απερίφθη. 231 Ολενίτσκα. Λίγη. Απερίφθη. Ξεκινάει η ψηφοφορία 232. Ξεκινάει λίγη. Απερίφθη. 233. Ξεκινάει η ψηφοφορία 233. Λίγη η ψηφοφορία. Ενεκρίθη. 37 του εισηγητή. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 37. Λίγη. Ενεκρίθη. 235. Σμιτ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Η 235 απερίφθη. 236. Ξεκινάει η ψηφοφορία εάν ε, Λίγη. Ενεκρίθη. 237. Μαζί 237 και 239 ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Απερίφθη. 238. Ξεκινάει η ψηφοφορία στη 238. Λίγη. Ενεκρίθη. 230. Με συγχωρείτε. 240. Λέει ο πρόεδρος. Ξεκινάει η ψηφοφορία στη 240. Λίγη. Ενεκρίθη. Συμβιβαστική 18. Ξεκινάει η ψηφοφορία σχετικά με τη συμβιβαστική 18. Λίγη. Ενεκρίθη. 249. Κόστιντζερ. Ξεκινά η ψηφοφορία για 249. Λίγη. Απερίφθη. 248. Ντόρφμαν. Ξεκινά ψηφοφορία. Λίγη. Ενεκρίθη. 250. Λίγη. Ενεκρίθη. Τώρα ψηφίζουμε τη 251 Σμιτ. Ξεκινάει ψηφοφορία. Λίγη. ενεκρίθη. 252. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 252 Παπαστάμκος. Λίγη. Ενεκρίθη. 39 του εισηγητή. Λίγη. Ενεκρίθη. Στην επόμενη σελίδα ψηφίζουμε την τροπολογία 40 του εισηγητή. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Ενεκρίθη. Τώρα πάμε στην 257 Χέραντς και Ξεκινά λίγη. 257 Απερίφθη. 258. Ξεκινά. Ενεκρίθη. 41. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τη 41 του εισηγητή. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Για τη 41. Απερίφθη. 259. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Απερίφθη. 42. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τη 42. Λίγη. Εγκρίνεται. 260 ε, λεφόλ. Ξεκινά η ψηφοφορία. Λίγη. Απερίφθη. 61. Ξεκινάει η ψηφοφορία στη 261 με εγκίνες, εγκρίνεται. 43 πρέπει επίσης να ψηφιστεί. Ξεκινά ψηφοφορία, λίγη. Ενεκρίθη. Τώρα ψηφίζουμε την πρώτη τροπολογία του εισηγητή. Ε, ένα του εισηγητή. Ξεκινά, λίγη, εγκρίνεται. Είμαστε στα εκτιμώντας, 46 Ντόρφμαν. Σαν ψηφίστε όλοι. Λίγη εγκρίθηκε 47. Ξεκινάει η ψηφοφορία στις 47. Λίγη. Σαράντα οκτώ. Ξεκινά η ψηφοφορία για τις 48. Είμαστε όλοι θετικοί. 48 λοιπόν. Λίγη ψηφοφορία 48 η οποία νεκρήθη. 49. Ξεκινά η ψηφοφορία σχετικά με το εκτιμώντας 11 και την τροπολογία 49. Τώρα 2 σχετικά με το εκτιμώντας 13 του εισηγητή. Ψηφίσατε, εγκρίνετε. Τροπολογία 50. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 50. Ενεκρίθη. 51. Συμφωνείτε όλοι για την 51. Ωραία, συμφωνούμε όλοι και εγκρίνεται. 52. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 52, θετική, άρα ενεκρίθη. 53, όχι. Άρα 54 τροπολογία Λάιον Ξεκινά ψηφοφορία για την 54. Λίγη. Απερίφθη. Η 54 απερίφθη λοιπόν. Τρία. Τροπολογία 3 του εισηγητή. Ξεκινά. Λίγη. Ενεκρίθη. 4. Τροπολογία 4 του εισηγητή. Ξεκινάει η ψηφοφορία, λίγη, ενεκρίθη. 57. Όχι, 56. Ψηφίζουμε πρώτα την 56 Λάιον. Λίγη ενεκρίθη. 57. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Ενεκρίθη. Πέντε του εισηγητή. Ξεκινά. Λίγη. Ενεκρίθη. Έξι, Ξεκινά. Λίγη. Ενεκρίθη. Και τέλος επτά, Ξεκινά. Λίγη. Ενεκρίθη επτά. Τώρα ψηφίζουμε την 58 ντελόνζ. Λίγη. Απερίφθη. 59. Ξεκινά ψηφοφορία για την 59. Λίγη. Απερίφθη. 60 ξεκινά η τροπολογία για την 60. Λίγη για την 60. Γέγκλε. Απερίφθη. Και τώρα ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 19. Ξεκινά. Ενεκρίθη. Τώρα την τροπολογία 66 ξεκινά ψηφοφορία στην τελευταία σελίδα, λίγη σχετικά με την 66, ενεκρίθη. Τώρα ψηφίζουμε τις τροπολογίες 9 του εισηγητή. Ξεκινά, λίγη, ενεκρίθη, 10 του εισηγητή, ξεκίνησε ψηφοφορία. Κλείνει. 11. Ξεκινά. Λίγη. Ενεκρίθη. Τώρα ψηφίζουμε την νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίστε όλοι παρακαλώ. Λίγη. Εγκρίνεται. υπέρ 32 ε, ο κανείς ε, κατά και δύο αποχές. Τώρα ψηφίζουμε την ε, το νομοθετικό ψήφισμα. Εγκρίθηκε. Και τέλος ψηφίζουμε την απόφαση να δώσουμε εντολή ε, για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για μία συμφωνία σε πρώτη ε, ε, ανάγνωση. Ψηφίσατε όλοι, συμφωνούμε όλοι και εδώ. Τρεις μόνο ψήφοι κατά. Ωραία, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε την κυρία Γκαρσία Πέρες. θέλει το Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους ε, της Επιτροπής μας για τη συνεισφορά τους και ιδίω τους και εισηγητής των διαφόρων ομάδων με τους οποίους ε, μπορέσαμε να συνεργαστούμε με πολύ καλό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ και για την καλή διάθεση που επέδειξαν για να βρούμε ε, συμβιβασμούς που μας επιτρέπουν να έχουμε μια στεναρή θέση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά να ευχαριστήσω και τα μέλη της Γραμματείας και τους βοηθούς μου χωρίς τους οποίους δεν θα υπήρχε δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά που καταφέραμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε η Ρέτσε. Ένα λεπτό την προσοχή σας παρακαλώ. Μη φεύγετε. Έχουμε ένα τελευταίο σημείο και θα πρέπει να σας παρουσιάσω μία έκθεση αρκετά σημαντική. Υπάρχουν κάποια διαφιλονικούμενα ζητήματα πολύ σημαντικά. Είναι το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ε, λίγα λεπτά προσοχή ακόμα. Σημείο 7 λοιπόν, 8 ε, στην ημερήσια διάταξη που έχουμε εμεί, κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Είμαστε στον κανονισμό για την ενιαία κοινή οργάνωση αγορά. Κείμενο για ευθυγράμμιση. Θα περάσουμε λοιπόν στη συζήτηση για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών ε, ε κανονισμός ε, ε του 2007 και βάσει των άρθρων 290 και 291 της Συνθήκης της Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρέπει να γίνει ευθυγράμμιση και όπως ε, κάναμε και για τα προηγούμενα θέματα έχουμε τη διαδικασία αυτή η οποία αφορά ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, την κοινή οργάνωση αγοράς. Ίσως και το πιο περίπλοκο όλης της γεωργικής νομοθεσίας και επομένως δεν ήταν εύκολο να το επανεξετάσουμε ε, λόγω της συνθήκης. Στην έκθεση που σας προτείνω υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες στόχο έχουν να αντικαταστήσουν εκτελεστικές πράξεις με πράξεις κατεξουσιοδότηση. Και υπάρχουν και κάποιες πράξεις οι οποίες θέλουν να αντικατοπτρίζουν την διατύπωση που έχει ήδη συμφωνηθεί με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Το πιο ευαίσθητο σημείο όμως, και εδώ θα ήθελα την προσοχή σας, και το πιο πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο θα ήθελα να επισημάνω εδώ ως εισηγητής είναι το άρθρο 43 παράγραφος 3 της συνθήκης δηλαδή τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την πρόταση ευθυγράμμισης. Ενώ στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου η συνθήκη καθορίζει την νομοθετική διαδικασία που χρησιμοποιείται ως συνήθως σε θέματα γεωργίας, δηλαδή συναπόφαση στην οποία ε, αρχίζουμε και συνηθίζουμε. Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου υπάρχει μια παρέκκληση που επιτρέπει μόνο στο Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εγκρίνει μέτρα που αφορούν τον καθορισμό των τιμών, των δασμών, των επιδοτήσεων και των ε, ποσοτικών περιορισμών επειδή είναι παρέκκληση, το άρθρο 43 παράγραφος 3 θα πρέπει να ερμηνεύεται κατ' εμέ με πολύ περιορισμένο τρόπο για να μην περιορίσει τα νομοθετικά δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μας οδηγήσει και σε μια κατάσταση η οποία θα ήταν κατάσταση πριν τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η Επιτροπή όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της, χρησιμοποιεί την παράγραφο 3 του άρθρου 43 που επαναλαμβάνω αποκλείει εξ ολοκλήρου το Κοινοβούλιο από την νομοθετική διαδικασία για αρκετές περιπτώσεις, ε, για την υποχρεωτική επιδότηση για το βούτυρο, για την ε, ανακατανομή του τομέα της ζάχαρης, ε, για τις επιδοτήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στο γάλα εν γέννη. για τα προϊόντα που δίνονται για τα σχολεία, για τις επιδοτήσεις στον τομέα της γεωργίας. Σε οκτώ άρθρα της κοινή οργάνωσης αγοράς, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αποκλειστεί εξ ολοκλήρου το Κοινοβούλιο από τη διαδικασία λήψης απόφασης. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω εδώ και δεν θα ήθελα να ξεκινήσω διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εμείς είχαμε επισημάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή μου στον Επίτροπο Τσόλος και το ζήτημα και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Απριλίου παρουσίασε μια πρόταση κανονισμού μόνο του Συμβουλίου που θέλει να εφαρμόσει τους συγκεκριμένους τομείς της κοινή οργάνωσης αγοράς καθορίζοντας τους κανόνες και τα μέτρα για τον καθορισμό των τιμών και τα υπόλοιπα χωρίς να υπάρξει συμφωνία σε αυτό το κείμενο ευθυγράμμισης. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια παράκαμψη, θεσμική αγένεια αν θέλετε και αν το Συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση κανονισμού πριν από την ευθυγράμμιση για την κοινή οργάνωση αγοράς, πριν από τη διαπραγμάτευση λοιπόν για την ε, ε, κοινή οργάνωση αγοράς, ε, θα αποτελέσει σαφώς πάρα πολύ αρνητική ένδειξη και για τις αρχές της αγαστής ε, διοργανικής συνεργασίας ε, που χρησιμοποιούμε μέχρι τούδε. Ως εισηγητής λοιπόν θεώρησα ότι θα πρέπει να διαγραφούν όλες οι αναφορές στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 και να συμπεριληφθεί αυτό που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κανονισμό μόνο του Συμβουλίου. Και κατά αυτόν τον τρόπο οι διατάξεις θα είναι στη βασική πράξη και θα υπάρχει συγκεκριμένος ρόλος Κοινοβουλίου και Συμβουλίου χωρίς να αποκλείεται το Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω λοιπόν να μπορέσετε να υποστηρίξετε τη θέση μου, διότι η πρόθεσή μου είναι να ενισχύσω το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να επιτρέψω την πραγματική εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνα. Και ελπίζω να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε αυτόν τον κανονισμό το συντομότερο δυνατόν, διότι η ε, προσεχής ε, ουσιαστική μεταρρύθμιση της διαδικασίας της κοινής οργάνωσης ε, οργανωράς θα επιβαρυνθεί από ένα επιπλέον στοιχείο εάν ακόμα παραμείνει σε κρεμότητα το θέμα αυτό της κοινής οργάνωσης αγορής. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Να σας πω ότι υπάρχει και προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 23 Ιουνίου 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε 11 και 12 Ιουλίου στην Επιτροπή μας το ζήτημα. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Πρόκειται για ευαίσθητη κατάσταση. Το άρθρο 43 παράγραφος 3 και η χρήση του είναι ιδιαίτερα σημαντικά και να δώσω το λόγο σε όσους θέλουν να παρέμβουν. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ στον ε, Πρόεδρο και εφόσον είμαστε στο τέλος της ημερησίας διάτασης θα ήθελα να πω ε, εις ε, το μέλη της Επιτροπής ότι αυτά που είπε ε, σχετικά με το άρθρο 147 παράγραφος 3 ο πρόεδρος είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο διότι διαφορετικά θα αποδυναμωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας διότι τα δικαιώματα αυτά τα οποία μας χορηγούνται μέσω του άρθρου 143 παράγραφος 3 θα μας αφαιρεθούν είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει στο ΕΛΚ και συνάδει η άποψη που έχει διατυπωθεί με αυτήν του Προέδρου. Ε, θέλω λοιπόν να τονίσω και πάλι αυτό το σημαντικό θέμα, δηλαδή ε, το άρθρο 143.3 είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε διότι διαφορετικά δεν θα έχουμε τα δικαιώματα συναποφάσεως. Ευχαριστώ τον κύριο Γιάρ για την παρέμβασή του, διότι δεν ξέρω αν ήμουν αρκετά σαφή στην παρουσίασή μου. Πρόκειται για οπισθοδρόμηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει κανονισμό στο Συμβούλιο βάσει του άρθρου 43.3 αποκλείοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έχει ήδη προτείνει. Και αυτό σημαίνει ότι οπισθοχωρούμε σε σχέση με τη Λισαβόνα. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή, ε, θεωρούμε ότι αυτή είναι περιοριστική ερμηνεία και ότι η συγκεκριμένη παρέκκληση αφορούσε μόνο συγκεκριμένες πράξεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια βήματα προ τα πίσω. Υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει το λόγο. Αν δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει από πλευρά Ευρωβουλευτό, θα ήθελα να δώσω το, ρόλο, το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εδώ ο κύριο Πατσέκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Δεκάστρο για την έκθεσή σας, για αυτή την πρόταση της Επιτροπής για την ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο που η γενική προσέγγιση της Κομισιόν υποστηρίζεται από εσά κύριε Πρόεδρε Ντεκάστρο. Το Δεκέμβριο εγκρίθηκε από την Κομισιόν και από τότε έγιναν πολλά για να τυποποιηθεί η προσέγγιση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη συνθήκη για τις κανονιστικές και κατά εξουσιοδότηση πράξεις και θα υπάρξει πλήρης ευθυγράμμιση με τη νέα οδηγία για την επιτροπολογία. Επίσης εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες που κάνατε, πρόεδρε Μοντεκάστρο, για τη βελτίωση της ποιότητας και της διατύπωσης. Παρακαλώ μόνο για να υπάρξει μεγαλύτερη ευληψία του κειμένου να μην επαναλαμβάνονται οι παραπομπές που δεν χρειάζεται να αναφέρονται εκατοντάδες φορές. Αλλά αυτό είναι τεχνικό θέμα. Επίσης συμφωνώ, Πρόεδρε, ότι ο στόχος και το εύρος για τις ε, πράξεις αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να εφαρμόζονται στις κατάλληλες περιπτώσεις. Και εδώ δεχόμαστε τις πρωτοπολογίες που βελτιώνουν το κείμενο, όχι όμως εκείνες που του αφαιρούν την ισορροπία μεταξύ των δύο τύπων πράξεων. Η ουσία είναι κάτι που το καταλαβαίνω αυτόν που είπατε για την ευθυγράμμιση αυτή κάναμε και παραπομπές στο άρθρο 43.3 και κάναμε και χωριστή πρόταση όπως είπατε και εσείς για το 43.3 της συνθήκης που προβλέπει με μονομένη δράση του Συμβουλίου με βάση πρόταση της Κομισιόν. Αλλά αυτό μόνο για ένα περιορισμένο αριθμό θεμάτων. Κατανοώ, Πρόεδρε, ότι είναι λεπτό για σας θέμα για το Κοινοβούλιο και προτείνετε στην έκθεσή σας οι ρήτρες του 43-3 να επαναληφθούν στο βασικό αυτό κανονισμό και με τις ποσότητες των θεμάτων. Θα ήθελα όμως να σας τονίσω ότι αυτό θα άφηνε κενό περιεχομένου το 43.3. Η συνθήκη αφορά βασικά και το 43.2 που είναι η βάση αλλά και την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιπτώσεων για, με το 43.3 και θα θέλαμε και οι δύο αυτές περιπτώσεις να καλύπτονται. Σας υπενθυμίζω εκ νέου ότι για μας δεν υπάρχει θέμα να εξαιρεθεί το Κοινοβούλιο από τη συμπερίληψη στη λήψη αποφάσεων για τα βασικά θέματα για το οποίο είναι αρμόδιο. Τέλος, συμφωνώ με την πρότασή σας ότι είναι επίγον να εγκριθεί αυτή η νέα οδηγία για να μην επιβαρυνθεί αχρίαστα και καθυστερήσει η συζήτηση για την ΚΑΠ και άλλες πράξη σε κάτι εξουσιοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πατσέκο. Ε, να ευχαριστήσω μόνο και να πω ότι το, η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά τι ακριβώς ε, γίνεται σε θέμα εφαρμογής του συγκεκριμένου κανονισμού και ελπίζω αυτή η προσέγγιση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτροπής ε, να ε, είναι αυτή που επιθυμεί και το Συμβούλιο και να συμφωνήσουμε και να έχουμε για το 43-3 μόνο τις απλοκλειστικές περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Αλλιώς ελοχεύει ο κίνδυνος να αποκλειστεί το Κοινοβούλιο και αυτό θα ήταν απαράδεκτο από πλευρά μας. Ευχαριστώ τον Διευθυντή Πατσέκο. Ε, ευχαριστώ όλους εσάς. Ε, θεωρούμε λήξασα τη συνεδρίαση και 27 Ιουνίου να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε συνεδρίαση από τις 4 μέχρι και τις 6 και μισή για την έγκριση του πακέτου των γαλακτοκομικών. Ε, να είστε όλοι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο επανειδήν.